να ανοίξουμε τα αυτιά μας για να ακούσουμε αυτά που ε, θα μας πούν και να υπογράψουμε τη δήλωση 13-2009 ώστε και άνθρωποι από, την Ανατολική, από τα ανατολικά Σύρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ελευθερία έκθεση. Κυρία Ντόιλ.